από κοντά την κατάσταση και εν παραστή ανάγκη θα παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Επίτροπε Κάλλας. Και τώρα έχουμε έξι ψηφίσματα. Θα γίνει ψηφοφορία μετά από το θέμα. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη το θέμα της Ιεμένης, αντική ποινή εναντίον ανηλίκων ατόμων, ιδιαίτερα η περίπτωση του Μουχάμετ Ταχέρ Θαμπέτ Σαμούμ. Να πάρουν το λόγο καταρχάς ε, οι συγητές. Η συνάδελφος Σάκα έχει ένα λεπτό το λόγο. Εκείνοι που περιφρονούν κάπως τη βία της κυβερνήσεως τους ε, έχουν προβλήματα. Το είδαμε τι έγινε στην Τινησία, στην Αίγυπτο, το Ιράν, την Αλγερία, τον Μπαχρέιν και στην Ιεμένη. Η νέα γενιά θέλει ελπίδα να αντικαταστήσει τον κινησμό να αντικατασταθεί η φτώχεια, η δικαιοσύνη, να αντικαταστήσει την ατιμορρησία και ελευθερία του διαδικτύου, να αντικαταστήσει ε, τη φήμωση και έχουμε πολλέ επίδειε στην Ιεμένη όσον αφορά την ανεξαρτησία. Βοηθούνται πολλά να γίνουν για την ελευθερία των, του δικαστικού και να, όλοι να εκφράζονται ελεύθερα. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα ανησυχούμε λόγω του κλίματο φόβου που έχει ε, μέσω τη εκτέλεση των νέων. Παρά τη δέσμευση τη Ιεμένη συμμορφωθεί με τα αυτά που επιτάσσει η διεθνή κοινότητα και ότι έχει δεσμευτεί να μην εκτελεί ανηλίκους ε, σύμφωνα με τον ποινικό της κώδικα. Υπάρχει έλλειψη επαρκών μέσων για να καθοριστεί η ηλικία των κατηγορουμένων. Είναι δύσκολο λοιπόν να υπερασπιστούν οι κατηγορούμενοι τον εαυτό του. Καλούμε τον πρόεδρο τη Εμένη και τι αρχέ να σεβαστούν τουλάχιστον του νόμου Ιεμένη και τι δεσμεύσει που έχουν αναλάβει τι διεθνού κοινότητε και να σταματήσουν οι εκτελέσει των ανηλίκων. Επίση, τονίζουμε την ανάγκη που υπάρχει για μεταρρυθμίσει στην Ιεμένη, κάτι που ζητήσαν πάρα πολλοί ε, διαδηλωτέ στου δρόμου και θέλουμε οι συνθήκε διαβίωσή του και τα δικαιώματά του να βελτιωθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε στην αδελφέ Σάκε και τώρα ο συνάδελφος Μερζιά για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι αραβικές χώρες ε, συγκλονίζονται από λαϊκές εξεγέρσεις και ελπίζω ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί. Ε, μια πνοή ε, επανάστασης έχει λειτουργήσει στην περιοχή. Αυτές οι δικτατορίες ε, της περιοχής ε, έχουν την εξουσία με την ε, σιωπηρή συνένεση των δυτικών χωρών. Καθυστερήσαμε, καθυστερήσατε να κατανοήσετε τα, τι συνέβαινε σε αυτές τις χώρες και συνεχίζετε να το πράτετε. Χρειάστηκε να περιμένουμε τη Δευτέρα Φεβρουαρίου προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει ένα ψήφισμα για την Τινησία. Και σε αυτή τη σύνοδο ψηφίσαμε και μια, ένα ψήφισμα για τον Αίγυπτο. Ζητήσαμε και ένα ψήφισμα για την Αλγερία. Αυτό μας το αρνήθηκαν για μια ακόμα φορά όπως συμβαίνει εδώ και μήνες, τουλάχιστον όπως η συλλογική πλησοφία μόν με ύψιλον είδε έκλειναν τα μάτια στα τεκτονόμενα στην ε, την Ισία. Σήμερα αυτή τη στιγμή στο Ιράν, στη Λιβύη γίνονται, υπάρχουν διαμαρτυρίες ε, με τι χώρε αυτέ υπάρχει και μια συμφωνία εταιρική σχέση, αλλά και στον Μπαχρέιν, την Ιεμένη, για να μην αναφέρω παρά μόνο χώρε ε, τι οποίε γνωρίζουμε καλύτερα. Στην Ιεμένη, όπου ο πρόεδρο Αλή Αμπταλέ Σαλέ βρίσκεται στην εξουσία μόνο 33 χρόνια. Ιδού λοιπόν μια δημοκρατία. Φυσικά είναι πολύ καλύτερα από τα ό,τι συμβαίνουν στην ε, Λιβύη, διότι ο κ. Καντάφη είναι στην εξουσία εδώ και 42 χρόνια. Μα είπαν ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα ένα ψήφισμα για την Ιεμένη, δίχω να λάβουμε υπόψη τα, τι συμβαίνει στη χώρα αυτή. Άντρε και γυναίκε αγωνίζονται για την ελευθερία ε, του. Συγκρούσει ανάμεσα στου πολέμιου και τι προσεχθέ του καθεστώτο. Εκατοντάδε άτομα έχουν τραυματιστεί. Χθε στο Άντεν ένα νέο σκοτώθηκε από σφαίρε τη αστυνομία που άνοιξε πυρ για να διαλύσει μια συγκέντρωση. Αυτή τη στιγμή ε, Φοιτητέ του ΣΑΔΑ βρίσκονται στο, κλεισμένοι στο πανεπιστήμιο και εμεί παραμένουμε σιωπηροί. Παρατηρούμε ότι το, υπάρχει το ζήτημα επίση της θανατικής καταδίκης ε, για του νέου. Εγώ ήμουνα πάντα υπέρ της ε, κατάργησης της θανατικής ποινή. Θεωρώ ότι κάθε δημοκρατική χώρα που δεν μπορεί να ε, απαγορεύσει μια τέτοια τιμωρία δεν μπορεί να δίνει μαθήματα ακόμα και αν αυτή είναι η πρώτη, παγκόσμια δύναμη. Και ξέρουμε πως ε, αυτή τη στιγμή ε, και για ποιους λόγους ε, καταδικάζονται σε θάνατο πολύ ανήλικοι στην χώρα αυτή. Θέλετε λοιπόν ψηφίσουμε ένα ψήφισμα το οποίο αφορά μόνο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή τη θανατική ποινή, αλλά και στο οποίο στο ε- σημείο 7 αναφέρεται η ανάγκη να τα αριθμίσει στην Ιεμένη όπω το ζητούν οι πολυάριθμοι διαδηλωτέ που έχουν κατέληξει του δρόμου. Εμεί έχουμε καταθέσει τρει τροπολογίε για να επικαιροποιήσουμε αυτό το ψήφισμα και ελπίζω πω όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε ένα κείμενο που θα μας αντιπροσωπεύει. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πρέντα, ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καθησυχάσω. Ε, όπως είπαν, όπως μπορούν να διαπιστώσουν όλοι, συζητούμε όχι μόνο τη θανατική ποινή, αλλά και αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους της ε, Ιεμένης εδώ και μερικές μέρες τη στιγμή ψηφοφορία θα μπορούμε να δούμε και ποια είναι η τοποθέτηση τη ομάδα μα όσον αφορά αυτά τα θέματα. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο στόχο του ψηφίσματο στα κατεπήγοντα αφορά την εφαρμογή της θανατικής ποινή επί των ανηλίκων. Όπως γνωρίζετε για μας Ευρωπαίους θανατική ποινή είναι μια βαρβαρότητα παράδεκτη και είναι ακόμα πιο φρικτή όσον αφορά την εκτέλεση ανηλίκων. Η θανατική ποινή για τους ανήλικους αντιτίθεται και στην ίδια την ομοθεσία της Ιεμένης. Όμως οι αρχές της χώρας αυτής εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυτή την πρακτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, στην Πρέντα. Και τώρα, 1,5 λεπτό, ο την σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα των κατεπηγόντων είναι ε, αυτό πάρα πολύ σημαντικό και να καλέσω τον Πρόεδρο τον Ιεμένη να αναβάλει την ε, ε θανατική ποινή, την ε, εκτέλεση του Μπετσάμου και άλλων ε, ανηλίκων όπως τον Αλή Αμπτούλα. Ωστόσο πιστεύω όπως αναφέρθηκε ότι θα ήταν ατυχές να χάσουμε την ευκαιρία αυτή για να θέσουμε κάποια από τα πιο βασικά και γενικότερα θέματα σε ό,τι αφορά τη χώρα αυτή. Και γι' αυτό θα ήθελα το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε να αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι η Εμένη όπως ε, η Αιγυπτός και η Τινησία χαρακτηρίζεται από διαδηλώσει. Ε, ατόμων που ζητούν εκδημοκρατισμό του κράτους, ενώ πολλοί διαδηλωτές υπέστησαν επιθέσεις και συλλήφθησαν. Αυτή ήταν η πρώτη μας ε, τροπολογία. Αλλά και δεύτερον ότι εκφράζει τη λύπη του για τα προβλήματα της Ιεμένης και θέλει να αποτραπεί η κλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης και τρίτη τροπολογία ότι εκφράζει την αλληλεγγύη αλληλεγγύη του προς τους διαδηλωτές που ζητούν βελτίωση του βιωτικού τους επίπεδου και καλωσορίζει την ε, δήλωση του Προέδρου ότι θα αποσυρθεί από την εξουσία του 2013 και ζητά να απελευθερωθούν οι διαδηλωτές που ειρηνικά διαδήλωση. Αν ε, συμπεριληφθούν αυτές οι τροπολογίες, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλό το ψήφισμα. Ευχαριστώ και τώρα η συνάδελφος Κρέτου, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξή. Η θανατική ποινή είναι απάνθρωπη ποινή, η οποία αντιστοιχώ εξακολουθεί να επιβάλλεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέφθινε έκκληση και ζήτησε να ε, καταργηθεί η θανατική ποινή όπου υπάρχει η εκτέλεση. Είναι ακόμα πιο φρικτή εφόσον πρόκειται για ανηλίκους, πρόκειται για ε, εγκλήματα τα οποία διέπραξαν ανήλικοι, παιδιά. Η Εμένη έχει υπογράψει τις σχετικές συνθήκες και το ποινικό δίκαιο της χώρας αυτής προβλέπει εμ, απαγόρευση της θανατικής ποινής για ανηλίκους. Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής ηλικία καθώς δεν υπάρχει επιστοποιητικό γέννησης και η συνέπεια είναι να μην εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο η θανατική καταδίκη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση στην Ιεμένη. Οι αρχέ παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλοί κλείνονται στη φυλακή. Είναι διακριτική η μεταχείριση κατά των γυναικών. Δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία, στη δημόσια ζωή. Δεν είναι αμερόληπτη η απόδοση της δικαιοσύνης. Οι διαμαρτυρίες υποδεικνύουν τις κοινωνικο-οικονομικές ε, πτυχές, αλλά υπάρχει και έκκληση για περισσότερη δικαιοσύνη στην Ιεμένη. Ευχαριστώ, συναδελφέ Κρετού. Και τώρα συνάδελφο Τάνοκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, συμμετέχει στα Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Εθνή Συμφωνία για τα Πολιτικά και ε, Δικαιώματα που απαγορεύουν την εκτέλεση των ανηλίκων κατηγορμένα. Αυτοί που καταδικασμένοι για εγκλήματα που ε, ε, έχουν διαπραχθεί όταν είναι κάτω από 18. Ο Μοχάμεν Σαμούν που πρόκειται να εκτελεστεί και που περιμένουν και πολλοί άλλοι ενήλικοι εκτελεστών άλλωστε, αυτό είναι ντροπή εναντί του διεθνούς δικαίου. Αλλά η εφαρμογή των πολιτικών λέγοντα ότι δεν έχουν επιστοποιητικό γέννηση σωστό και υπάρχει αμφιβολία για την ηλικία του, ευθυγραμμίζεται η Εμένη με τη θεοκρατία την ομή του Ιράν. Όμω η διαφορά μεταξύ των χωρών είναι ότι η Εμένη παίρνει τεράστια βοήθεια από τη Δύση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκριζώσει του τρομοκράτε τη Αλκάιντα. Ενώ το Ιράν είναι ένα διεθνή ε, περιθωριακός Λοιπόν, θα πρέπει να παρατηρήσουμε έκθεση στον Αλή Αμπτού Ασάλε, τον πρόεδρο, να, να ζητήσουμε ε, να δείξει φιλεφταχνία όσον αφορά αυτή την εκτέλεση. Εφόσον θα φύγει από τη θέση, το πρόεδρο Σαλέ έχει πραγματική ευκαιρία να αφήσει ένα αποτύπωμα, μια κληρονομιά θετική ε, που έχει υποστεί ε, την τρομοκρατία επί τόσα χρόνια και ονειρεύεται τώρα για ένα δημοκρατικό μέλλον. Ευχαριστώ, συνάδελφε Τάνοκ. Και τώρα να σας παρακαλέσω, συνάδελφε Τάνοκ, Συνάδελφε Τάνοκ, να σας παρακαλέσω στο μέλλον να μιλάτε λίγο, να διαβάζετε λίγο ε, πιο σιγά. Ίσως αν θέλετε να κατανοεί ο κόσμος αυτά που λέτε όχι μόνο στα αγγλικά, μην γράφετε τόσο πολλά στο κείμενό σας γιατί δυσκολεύετε πάρα πολύ τους ε, διερμηνείς. Και τώρα, εξ ονόματος των ομάδων, ο κύριος Κατσμάρεκ ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 1991 στην Ιεμένη οι εκτελέσεις ανηλίκων απαγορεύτηκαν. Αλλά από το 1994 και μετά η απαγόρευση αυτή αφορά τα άτομα κάτω των 18. Ωστόσο δεν γίνεται σεβαστή αυτή η απαγόρευση. Πολλά άτομα όπως αναφέρθηκαν δεν έχουν επίσημα έγγραφα που να πιστοποιούν την ηλικία τους, αλλά υπάρχουν και άλλα ανασχετικά φαινόμενα. Τα όπλα στην Ιεμένη είναι πιο πολλά στον αριθμό από ότι οι κάτοικοι της Ιεμένης. Οι συγκρούσεις αποτελούν καθημερινή ρουτίνα και συχνά συμμετέχουν παιδιά σε αυτές. Ο κόσμος λέει ότι αν είσαι αρκετά μεγάλος για να κουβαλάς μαζί σου μαχαίρι, μπορείς και να πολεμήσεις. Το να βλέπει κανείς ένα παιδί, έναν έφηβο με ένα καλάσνικοφ δεν είναι περίεργο θέαμα. Η κοινωνία της Ιεμένης είναι πολύ νέα στην ηλικία. Το 50% είναι κάτω το 18% και πολλοί προσπαθούν να στρατολογήσουν ε, τους νέους. Θα πρέπει και αυτό να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ στην Κασμάρεκ. Η κυρία Γετεμέκη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, σε 58 χώρες υπάρχει ακόμα θανατική ποινή και μία από τις χώρες αυτές είναι και η Εμένη. Η ομάδα μου καταδικάζει αυτή την ποινή εν γέννη και τη σχεδιαζόμενη εκτέλεση του Μοχάμετ Αμπέτ Σαμούν ιδιαίτερα. Θέλουμε να θυμίσουμε στην κυβέρνηση της Ιεμένης ότι έχει διεθνείς διασμεύσεις. Έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Πολιτικά Δικαιώματα και οι δύο συμβάσει απαγορεύουν την εκτέλεση ανθρώπων κάτω των 18. Κύριε Πρόεδρε, τη Δευτέρα η Διεθνή Αμνηστία ανέφερε τις δράσεις των δυνάμεων ασφαλεία τη Ιεμένης. Σύμφωνα με την αμνηστία, οι δυνάμεις ασφαλείας έδιραν διαδηλωτέ με ξύλα και χρησιμοποίησαν και ηλεκτρικά ραβδιά για να τους δώσαν ηλεκτροσόκ. Καταδικάζει αυτές τις δράσεις βίας η ομάδα μου και παροτρύνει την κυβέρνηση της Ιεμένης να παρετηθεί της χρήσης βίας κατά του λαού της Ιεμένης. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Γετεμέκη. Και τώρα ο συνάδελφος Τζανέσκι για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπόσχομαι πως ε, δεν πρόκειται να αναγνώσω την ε, λόγο μου θα, και θα μιλήσω αργά. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που λαμβάνω το λόγο μετά από την πρώην ε, Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας. Έχουμε μια μινιμαριστική προσέγγιση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε, κάνουμε έκκληση προς τις αρχές να απαγορεύσουν την θανατική ποινή για τους νέους. Εγώ είμαι κατά της θανατικής ποινής, μόλον ότι γνωρίζω ότι στην αίθουσα αυτή έρχονται και κάποια άτομα τα οποία είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Είτε Εγώ είμαι κατά, είτε πρόκειται για ανηλίκους, είτε για ενηλίκους. Αλλά θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί εάν μιλήσουμε με μία φωνή προς τις αρχές της Ιεμένης. Ο πρόεδρος της εν λόγω χώρας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το, το δικαίωμα που δίνει ε, ο Σύνταγμα για επίοικια. Ευχαριστώ. Ο πως Πάσκα ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, τα δικαιώματα των παιδιών και οι άλλες ε, συνθήκες είναι συνθήκες που έχει υποσχεθεί να αποδεχτεί η κυβέρνηση της Ιεμένης και βάσει των ε, εγγράφων αυτών, των συνθήκων αυτών, ε, απαγορεύεται η θαντική ποινή. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να λαμβάνει τέτοιες νόμιμες αποφάσεις η Ιεμένη, αντιβαίνοντας στις συνθήκες αυτές. Οι θανατικές ε, καταδίκες αυτές δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι θέλει να σεβαστεί τις δημοκρατικές αρχές. Δεν μπορεί λοιπόν να εφαρμόσει τέτοιες θαντικές καταδίκες. Αυτό το γεγονός θα πρέπει λοιπόν σήμερα να το τονίσουμε στην ε, κυβέρνηση της Ιεμένης. Ευχαριστώ, συνάδελφε Πάσκα και τώρα 1,5 λεπτό ο, ο συνάδελφος Σέγκεντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ασφαλώς θεωρώ ότι είναι σημαντικό να καταδικάσουμε δικτάτορες και δικτατορικά καθεστώτα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και γενικότερα την Ιεμένη να οδεύσει προς τον εκδημοκρατισμό. Τώρα που το θέμα της Ιεμένης έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη, δεν είναι όμως ε, δικό μας καθήκον να καθορίσουμε και να αποφασίσουμε ε, επί τη υπόθεση της Ιεμένη. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα και είναι ασαφέ, καθότι δεν, γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες του δικαστικού συστήματος, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι ηλικία είχε το άτομο αυτό όταν ε, διέπραξε τα εγκλήματα τα οποία υποτίθεται ότι διέπραξε. Δεν ξέρουμε αν ήταν ενήλικος ή ανήλικο στην εποχή εκείνη. Δεν υπάρχει καν πιστοποιητικό γέννησή του. Τα χαρτιά, τα πιστοποιητικά ε, του σχολείου που παρουσιάστηκαν δεν ξέρουμε αν είναι πρωτότυπα ή όχι. Δεν μιλάμε για ένα πτέσμα, μιλάμε για φόνο. Διαπράχτησε φόνος. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πρωτού αποφανθούμε από αυτού. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, υπάρχουν σοβαρά εγκλήματα στα οποία δικαιολογείται η εφαρμογή της θανατικής καταδίκης. Ναι. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Σέγκετη. Και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, η συνάδελφος Εσάγια έχει καταρχάς το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση αυτή του Θαμπέτ Σαμούμου. Υπάρχουν ε, μια δεκαριά άτομα τα οποία περιμένουν τη σειρά τους για εκτέλεση θανατικής ποινής. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δεν έχουν πιστοποιητικά γέννηση και δεν γνωρίζουμε κατά πόσο πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους. Ως εκ τούτου χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πως η ΕΜΕΝΗ έχει επικυρώσει κάποιες διεθνείς συμβάσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των ανηλίκων συμβάσεις οι οποίες ε, αναφέρουν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η θανατική ποινή σε ανηλίκους. Η θανατική ποινή λοιπόν για έναν ανήλικο παραβιάζει ακόμα και τον ποινικό κώδικα της Ιεμένης. Και όχι μόνο, αλλά και τον διεθνή ποινικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Μπασέσκου έχει ένα λεπτό το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η καταδίκη ενός παιδιού σε θαντική καταδίκη είναι πραγματικά απαράδεκτη, ιδιαίτερα στο σημερινό κόσμο. Αυτή η πρακτική όμω έχει γίνει συνήθεια. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνώ με τις αρχές τη Ιεμένη σε ό,τι αφορά την συνέχιση της εφαρμογής της καταδίκης της θαντική. Οι αποφάσεις της κυβερνήσεω ε, αντιβαίνουν στι διεθνεί συνθήκε και στην ομοθεσία της ίδιας της χώρας που δεν επιτρέπει την καταδίκη ανηλίκων. Επιπλέον δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι το άτομο αυτό. Είναι πραγματικά λυπηρή αυτή η εικόνα που βλέπουμε στην Ιεμένη ως ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως ε, πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη ζωή πρόκειται για ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει τα παιδιά να προστατεύονται. Και θέλω να απευθύνω έκκληση προ την ύπατη εκπρόσωπο για να το θέσει το θέμα αυτό προ τον ηγεμένη και να θεθεί τέλο στι εκτελέσει αυτέ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μπασέσκου. Και τώρα η κυρία Μάκοβεϊ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πιθανότατα ο Αλή Αμπντούλ Σαμουν ήταν ανήλικος όταν ε, και οι δύο που κατηγορούνται ήταν ανήλικοι όταν διαπράξαν τα εγκλήματα δέχτηκαν αυτή την ποινή εδώ και χρόνια και αυτές οι ποινές ίσως ε, μπορεί να εκτελεστούν οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει μια ψυχολογική ε, πίεση τεράστια και ήδη ήταν απάνθρωποι η μεταχείρισή τους ζητούμε λοιπόν από τις αρχές να μην εκτελέσουν αυτούς τους ανθρώπους και οι δύο δεν μπορούν να αποδείξουν ότι ήταν κάτω των 18 ετών διότι δεν έχουν πιστοποιητικό γέννησης. Η απόκτηση των πιστοποιητικών είναι σοβαρό πρόβλημα στην Ιεμένη, όπου μόνο το 22% των γεννήσεων καταχωρούνται επίσημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ε, UNICEF. Ίσως ένα τμήμα των πόρων που διαθέτουμε στην Ιεμένη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επιληθεί το λόγο πρόβλημα. Η συζήτηση γύρω από αυτή την υπόθεση θα πρέπει να οδηγήσει στο εξή. Εκατοντάδες άτομα που είναι καταδικασμένοι σε θάνατο θα πρέπει τελικά να μην καταδικαστούν στο θάνατο, να αλλάξει η ποινή τους. Θέλω να το θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητήσεις με την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μακοβέη. Και τώρα η διαδικασία κατσδιάει και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συνάδελφο του Χόνσταϊν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είτε πρόκειται για ανηλίκους είτε για ανηλίκους. Η ανθρώπινη η καταδίκη σε θάνατο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε πιο επισταμένα. Έχουμε ένα κώδικα τεντολογίας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προωθηθεί και σε άλλες χώρες όπου έχουμε και διατηρούμε οικονομικές σχέσεις. Δυστυχώς στην Ευρώπη Υπάρχουν χώρες που ακόμα εφαρμόζουν την θανατική καταδίκη. Αυτά που συμβαίνουν στην Ιεμένη σημαίνουν ότι θα πρέπει να απευθύνουμε κατεπίγουσα έκκληση προς την κυβέρνηση της χώρας για να σταματήσουν αυτές οι ε, απάνθρωπες πρακτικές. Και να σας υπενθυμίσω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα ε, ποινείται στις φυλακές και οι πιο πολλοί από αυτούς είναι ανήλικοι. Θα πρέπει πιο στο να συνεργαστούμε επίσης με την Διεθνή Αμνηστία. Και με το Ίδρυμα του Ελσίνκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να ακουστεί επιτέλους η φωνή μας. Ευχαριστώ, συνάδελφε του Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Όμπερ Μάιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. είναι πραγματικά φρέχτες πρακτικές θανατικής καταδίκης ανηλίκων. Είναι παράνομες ε, οι πρακτικές αυτές της ε, Ιεμένης, γιατί η Ιεμένη έχει υπογράψει τη συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού και το άρθρο 37 ε, ορίζει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν θανατικές καταδίκες σε άτομα που είναι κατά των 18. Αναφέρεται ως δικαιολογία ότι δεν μπορεί να οριστεί η ηλικία του κατηγορούμενου, αλλά Στη Σομαλία, για παράδειγμα, τα δικαστηρία Σαρία ε, επιβάλλουν τη θανατική καταδίκη σε νέου Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΟΗΕ θα πρέπει να δράσει γρήγορα και με μεγάλη αποφασιστικότητα για να επιβληθεί το διεθνέ δίκαιο με όλε τι σχετικέ κυρώσει. Καλό είναι να μιλάμε κυρίε και κύριοι, αλλά θεωρώ ότι τα πολιτικά και οικονομικά επιχειρήματα νομίζω είναι πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα, στο τέλος της διαδικασίας κάτω στο ο συνάδελφος Σιλβέστης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ενώ εμείς συζητάμε, εκατοντάδες κρατούμενοι περιμένουν ε, να εκτελεστούν στις ε, φυλακές της Ιεμένης. Νομίζω ότι θα χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η συνεχής παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να βλέπει την Ευρώπη απούσα και σιωπούσα. Με την Ιεμένη έχουμε σχέσεις και οικονομικής φύσης, κάτι το οποίο χρειάζεται να μας ε, κάνει να σκεφτούμε περισσότερο το μέλλον αυτών των σχέσεων. Είναι προφανές ε, πως στην Ευρώπη το ζήτημα της ε, κατάργησης της θανατικής ποινής είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιβληθεί και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να χρησιμεύσει για την βελτίωση των συνθήκων Ευχαριστώ, Στάλφε Σιλβέστρη. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Κάλλα. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις γραμμές για τη θανατική ποινή επί μακρόν ήταν δραστήρια στην καταπολέμηση θανατικής ποινής και στην Ιεμένη και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε η θανατική ποινή ε, εκτελέσεις ανηλίκων λάβαναν χώρα πάντα στην Ιεμένη. Παλαιότερα όμως δεν γινόταν γνωστές και η κοινωνία των πολιτών δεν ήταν τόσο δραστηριοποιημένη. Λοιπόν, υπάρχει πρόγραμμα δικαιοσύνη υπέρ των ανηλίκων που χρηματοδοτείται από, τον, από τη UNICEF και από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο στο πρόβλημα. Εφαρμόστηκε και με διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με το Συμβούλιο για τη Μητρότητα και τα Παιδιά. Πώς έγινε η προσπάθεια ευαισθητοποίηση. Δεν αρκεί η ευαισθητοποίηση όμω. Θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια με δράσει. Σαν τελευταία γραμμή δράση, η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω κάνει διαβήματα για να σταματήσουν εκτελέσει. Δύο πρόσφατε περιπτώσει το Δεκέμβριο του 2004, Φαχουάρα Λίβα Αμπτούλα και τον Ιανουάριο του 2011 για τον Σαμούν. Και στις δύο περιπτώσεις η εκτέλεση πάγωσε μετά από παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά αφορά την ηλικία τους. Ο Μοχάμετ Αμπέτ Ταχέρ Σαμούν το θέμα αυτό ξανατέθη στο προσκήνιο την περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται ότι ίσω τελικά ε, αλλάξει, δοθεί χάρη από τον πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNICEF ήρθαν σε επαφή με τον πρόεδρο Σαλέ και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τη ΣΑΝΑ η εκτέλεση ξανά έχει σταματήσει. Δεσμεύεται από διεθνείς υποχρεώσεις η Εμένη δεσμεύεται και από την νομοθεσία της για δικαιοσύνη επί ανηλίκων και από τον ποινικό της κώδικα δεσμεύεται να μην εκτελεί τους ανηλίκους. Γιατί περιμένουν εκτέλεση οι ανήλικοι λόγω ελλείψεως δυνατότητας καθορισμού της ηλικία βασικά. Μαζί με την UNICEF πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ιεμένη να δημιουργήσει, να αποκτήσει εμπειρία, γνώση σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Ενδιάμεσα, μεσοπρόθεσμα, θα ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα που θα επανεξετάσει το θέμα τη ηλικία. Θα έχουμε σαν στόχο την υποστήριξη της δυνατότητας που θα έχουν οι δικηγόροι να υπερασπίζονται στο δικαστήριο του ανήλικους. Και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τη δημιουργία μια μιας που θα καταχωρεί, θα καταρτήσει μητρώα ηλικία. Θα πρέπει να διτεχθούν όλα τα μέσα για να βρεθεί λύση. Η κυβέρνηση εμένη ε, ήταν δεκτική στα διαβήματά μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να του βοηθήσει και τώρα και στο μέλλον. Ούτω ώστε να σταματήσει η εφαρμογή θανατική ποινή. Ευχαριστώ την προσοχή σα. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Κάλλας και τώρα ε, έχουμε έξι προτάσεις ψηφισμάτων και οι ψηφοφορίε θα γίνουν με το τελευταίο θέμα. Επόμενο ζήτημα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα